Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Φαντάζομαι ότι έχετε φέρει όλοι μαζί σας τις ε, ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, εγκρίνουμε την ημερήσια μας διάταξη. Σημείο 2. Ε, να μεταδίδεται, στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μας. Έχουμε διερμηνία σε 20 γλώσσες, με εξαίρεση τσεχικά, μαλτέζικα, σλοβακικά και κελτικά, ιρλανδικά. Ε, ε, η κυρία Χόιμπουχ κάλεσε μια ομάδα κινηματογραφική στη συνεδρίαση γιατί γυρίζουν ένα ντοκιμαντέρ. Επίσης, ε, και ο κύριος Δενανό έχει καλέσει κάποιους δημοσιογράφους από ένα τοπικό τηλεοπτικό κανάλι. Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών της σα διάταξης της 12ης Μαρτίου, 19ης και 20ης Μαρτίου, 12ης Απριλίου και 23 και 23 και 24 Απριλίου. Ε, βάσει διαδικασία, αν δεν υποβληθούν παρατηρήσει μέχρι το τέλο συνεδρίαση, ε, θεωρούνται ω εγκεκριμένα τα πρακτικά. Και περνάμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σημείο πρώτο προ ψηφοφορία, οι ενοποιημένε στατιστικέ γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η συγκεκριά μα είναι η κυρία Μαρία Γαβριέλα Ζωανά. Ε, πρόκειται για την ε, προκτακτική συνεργασία μετά τις διοργανικές διαπραγματεύσεις. Τον Απρίλιο, στη συνεδρία της Επιτροπής, η συγκήτριά μας, η κυρία Ζωανά, μας ενημέρωσε για την προσωρινή συμφωνία με το Συμβούλιο στο θέμα των ενοποιημένων στατιστικών για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ε, και το σχετικό κανονισμό. Ε, αυτό επιτέθηκε στο τρίτο τριμερή διάλογο που έγινε στις 11 Απριλίου. Δυστυχώς υπάρχει ένα πρόβλημα με τον ήχο. Οπότε ε, έχουμε αυτή την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε και από την Κορεπέρ στις 8 Μαΐου. Δεν ξέρω αν η συγκεκριά μας έχει να προσθέσει κάτι. Παρακαλώ. Όπως είπα και στην ε, προηγούμενη συνεδρίαση, είχαμε τρεις ε, συναντήσεις ε, τον τριμερή διάλογο. Καταλήξαμε τελικά σε μια συμφωνία και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν. Ευχαριστώ. Ωραία, τότε ας περάσουμε στην ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία, γίνεται άπαξ ε, ψηφοφορία για το θέμα αυτό. Ψηφίσατε όλοι. Λίγο ακόμη περιμένουμε. Μια και είναι η πρώτη ψηφοφορία για να συνηθίσουμε. Εντάξει, τέλος ψηφοφορίας. Gratulujemy pani poseł. Ωραία, εγκρίνεται, οπότε περνάμε στη συνέχεια. Περνάμε επίσης στο δεύτερο τώρα σημείο, στο σημείο 5, το μέλλον της γεωργίας και των τροφίμων. Είναι η δική μας απάντηση στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μάλιστα χαίρομαι γιατί καταφέραμε σχετικά γρήγορα να καταρτήσουμε τη δική μας ε, έκθεση ώστε να περάσει γρήγορα στην Ολομέλεια πριν ε, υποβάλει την νομοθετική της πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί εκεί στα τέλη Μαΐου ή αρχές Ιουνίου θα υποβληθούν οι σχετικές νομοθετικές προτάσεις για την ΚΑΠ μετά το 2020. Θέλαμε λοιπόν να έχει κάποια βαρύτητα και δική μας γνώμη και γι' αυτό κρίναμε σκόπιμο να την ε, υποβάλουμε υποβάλλουμε εγκαίρως. Γνωμοδοτήσεις έδωσαν οι Επιτροπές Περιβάλλοντος Προϋπολογισμών Διεθνούς Εμπορίου, Ανάπτυξης και Ελέγχου Προϋπολογισμού Διαπιστολής και μάλιστα ο ενορχιστρωτής όλης αυτής της, ο διευθυντής ορχήστρας μάλλον όλης αυτής της διαδικασίας είναι ο εισηγητής μας, ο κύριος Ντόρφμαν, στον οποίο θα δώσω και το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Όπως ε, ήδη αναφέρατε, ε, αυτή την έκθεση την προετοιμάσαμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα γιατί ο στόχος μας ήταν ε, να δημοσιευτεί, να κατατεθεί η έκθεση αυτή πριν από τη δημοσίευση των νομοθετικών προτάσεων. Ελπίζουμε λοιπόν να κατορθώσουμε στην επόμενη Ολομέλεια στο Στρασβούργο να μπορέσουμε να ψηφίσουμε επί της έκθεσης αυτής. Και όλα αυτά τα καταφέραμε γιατί εργαστήκαμε επικοδομητικά. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω το σκιώδη συγητή και τους συγητέ των άλλων επιτροπών. Τους ευχαριστώ όλους ε, θερμότατα γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η επικοδομητική εργασία δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ολοκληρώσει εργασίες μας σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και ευχαριστώ και τους συνεργάτες γραμματείας, τους ε, οποίους πιέσαμε ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, γιατί η όλη δουλειά ήταν πάρα πολύ έντονη. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντέση το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το Ηράκλειο έργο, να ευχαριστήσω και τους σκιώδη εισηγητέ και τους συνεργάτες. Προχωρήσαμε πολύ γρήγορα, ευχαριστούμε γι' αυτό, ευχαριστούμε για την κατάρτιση του καταλόγου ψηφοφορίας. Έχω μόνο μία ε, παράκληση. Η τροπολογία 756 που περιλαμβάνεται στην σημαντική πρόταση 14 να ψηφιστεί ξεχωριστά. Γιατί βεβαίως αν υπάρχουν τόσες πολλές ε, τροπολογίες Μπορεί να συμβεί κάποια συμβαστική έκθεση να χαθεί, κάπου να χαθεί, να μην ζητήσει σημασία. Γι' αυτό θα ήθελα να ψηφιστεί ξεχωριστά η 14 συμβαστική πρόταση. Ο κύριος Αρντά. Ευχαριστώ. Έλα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους ε, σκιώδεις εισηγητές και όπως ε, και ο κύριος Ντες έχω και εγώ μια παράκληση σας παρακαλώ να βγει η 429 η τροπολογία από την συμβιβαστική πρόταση. Μιλάμε για την άρδευση εκεί. Στα κράτη-μέλη στα οποία η έκταση αυτή δεν φτάνει τον μέσω όρο της Ένωσης. Ε, αυτό είχε υποβληθεί από τους συναδέλφους Ικρίνσκι, Καλινόφσκι, Ντόρφμαν, ε, και Νέκοφ. Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ σημαντική τροπολογία. Ε, δεν την βλέπω λοιπόν και σας παρακαλώ να ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον κύριο Ντόρφμαν, για το πολύ αξιόλογο άρτιο έργο του. Συμφωνώ με τον κύριο Ντες και ευχαριστώ και τους κοιόδης εισηγητές για τη συνεργασία. Θα ήθελα εν ώψη της ψηφοφορίας να διαρωτηθούμε. Μήπως έχουμε την αίσθηση ότι παίζουμε το ρόλο του χρήσιμου χαζού, του χρήσιμου ηλιθίου. Γιατί στις 29 θα ψηφίσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, στην, ε, συγγνώμη, στην ε, Ολομέλεια. Ε, ενώ ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιτρέψει κάποιες διαρροές για τις νομοθετικές προτάσεις και δεν νομίζω ότι είναι σωστό και δημοκρατικό να παίζουμε εμείς το ρόλο του ωφέλιμου ηλιθίου. Γιατί αυτή την αίσθηση έχω. Νομίζω ότι θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει πιο σοβαρά το Κοινοβούλιο και το έργο του και να μην μας ε, περιγελά έτσι. Έχουμε ξοδέψει τόσο χρόνο για την έκθεση αυτή και νομίζω ότι εν ώψη και του μέλλοντος της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής ε, άκουσε περισσότερου σεβασμού εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η όλη διαδικασία και φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ας μην ανοίξουμε τώρα παρακαλώ συζήτηση. Δεν χρειάζεται όλοι να λάβετε το λόγο εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Γιατί έτσι θα παρατείνουμε ε, τη συζήτηση. Φαντάζομαι ο κύριος Ανδρία είχε ένα ζήτημα διαδικαστικό. Από εδώ και πέρα, μετά από τη δική μου παρέμβαση, ε, δεν χρειάζεται να λάβετε το λόγο διαδικαστικά ή να ευχαριστήσετε τον ίσιο γιατί τον έχουμε ευχαριστήσει. Ε, είναι όμως διαδικαστικό, μόνο για διαδικαστικά παρακαλώ από εδώ και πέρα, όχι απλώς για ευχαριστήσεις ή άλλα θέματα. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντόρφμαν και τους ε, σκιώδης συγητές. Ε, να σας βοηθήσω. Τι θέλετε. Λοιπόν, συζητήσαμε επί τη βάση επιχειρημάτων και όχι ιδεολογιών. Βεβαίως, ε, κύριε Ντες, πολλές από τις ε, πράσινες τροπολογίες πήγαιναν πιο πέρα από τον συμβασμό. Δεν ξέρω τώρα εάν πρέπει να επαναληφθούν αυτά εδώ πέρα. Εγώ προτείνω να παραμείνουμε στην ε, συμβιβαστική πρόταση και την διαδικασία ψηφοφορία που προτείνεται zawiera się... Κυρία Γκοσεύσκα, θέλετε οπωσδήποτε το λόγο. Δεν χρειάζεται να ανοίξουμε συζήτηση και όλοι να λαμβάνετε το λόγο για να ευχαριστείτε τον εισηγητή. Αυτό θα μα πάρει μισή ώρα να όλοι πρέπει να ευχαριστήσουμε ξεχωριστά τον εισηγητή. Σα ευχαριστώ. Εγώ έχω μια παρατήρηση για την 7η συμβαστική τροπολογία, για την ε, ε, άδικη εξίσωση των ενισχύσεων και τη λήψη υπόψη του κόστους παραγωγής. Είναι πραγματικά ρεαλιστικό αυτό το θέμα. Νομίζω ότι είναι ε, απάτη ότι, δεν, ότι, υποτίθεται ότι με τις ενισχύσεις. Και νομίζω ότι δεν πρέπει με βάση κάποιες περίεργες διατάξεις ουτοπικές και μη ρεαλιστικές να ισχυριζόμαστε κάτι τέτοιο. Ε, γιατί αναφέρονται κάποιες natural conditions, κάποιες ε, ε, φυσικές συνθήκες, υπεριστάσεις, το κόστος παραγωγής. Εγώ πιστεύω ότι οι ενισχύσεις θα πρέπει να εξισωθούν, στην ουσία όμως και όχι θεωρητικά, γιατί δεν υπάρχουν πια επιφυλάξει περιορισμοί, ούτε κανονιστικοί, ούτε λόγω των συνθήκων. Αντίθετα, θα πρέπει να εξισωθούν οι ενισχύσεις χωρίς όρους γιατί ποτέ οι γεωργοί δεν είχαν τις ίδιες ενισχύσεις και είναι άδικο ε, οι Πολωνοί γεωργοί για παράδειγμα να λαμβάνουν λιγότερες ενισχύσεις από τους Γερμανούς που είναι ε, γειτονική τους χώρα. Ανάλογα με το που είναι ως προς τα σύνορα, δηλαδή ο αγρότης να λαμβάνει διαφορετικές ε, ενισχύσεις. Αυτό είναι άδικο, γι' αυτό και δεν είμαστε σε θέση να υπερψηφίσουμε την έκθεση. Σας ευχαριστώ κύριε Ντόρφμαν, μήπως έχει, θέλετε το λόγο για να Απαντήσατε στην κυρία Γκοσεύσκα για αυτή την θέση που εξέφρασε ως προς την τροπολογία, ως προς την έκθεση. Κυρία Αγγιλέρα, εγώ θα ήθελα να πω ότι είχαμε ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή μας και πραγματικά επιτελέσαμε τιτάνιο έργο τις τελευταίες εβδομάδες. Και για να καταλήξουμε σε, αυτή την, σε αυτές τις λύσεις πραγματικά πασχίσαμε και μοχθήσαμε πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να προσθέτουμε τώρα διάφορε τροπολογίε, όσο σημαντικέ και αν είναι. Έχουμε καταλήξει συμβαστικέ τροπολογίε. Α ψηφίσουμε, ας ψηφίσουμε με βάση τον κατάλογο, χωρί αλλαγέ. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό τώρα τελευταία στιγμή να υποβάλουμε τροπολογίε, όπω έκανε ο κύριος Έρντοχ που έχει κάθε δίκιο αλλά είχαμε χρόνο για κάτι τέτοιο. Ήταν πολύ εντατικό το έργο που κάναμε ε, με στενή συνεργασία με τον εισηγητή, α αφήσουμε άθικτο τον κατάλογο ψηφοφορία με τι συμβαστικέ τροπολογίε. Όποιο διαφωνεί, α καταψηφίσει, εν πάση περιπτώσει. Ναι, αλλά α δώσουμε το λόγο στον εισηγητή μα, τον κύριο Ντόρφμαν, για να απαντήσει παρόλα αυτά. επί της αρχής δεν έχω κάποια αντίρρηση στο να ψηφίσουμε χωριστά αυτά τα δύο σημεία, αλλά ελπίζω μετά να συμφωνούν οι συνάδελφοι να πάνε στην ε, Ολομέλεια. Νομίζω ότι είναι και απλούστερο έτσι. Νομίζω ότι είναι καλύτερο από το να το κάνουμε τώρα εδώ τελευταία στιγμή. E, ο κύριος Δες νομίζω απέσυρε την τροπολογία του. Και ο κύριος Ερντός το ίδιο. Δεν θέλει να κάνει άλλο σχόλιο ο συγητής μας, ο κύριος Ντόρφμαν. Οι υπόλοιποι θα εκφέρουν τη γνώμη τους μέσω της ψήφου τους. Ευχαριστώ για την μέχρι τώρα συζήτηση και ας περάσουμε στην ψηφοφορία. Σας θέρμο παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια εμφανώς, κυρίως οι συντονιστές των ομάδων και οι σκιώδεις ηγητές. ε, κυρίως κοιτάω προς τα αριστερά γιατί από δεξιά είναι, κυρίως, είναι του ΕΛΚ. Ο κύριος ΕΚ, η τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας του κύριου ΕΚ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 1 του κύριου ΕΚ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Με μία ψηφοδιαφορά εγκρίνεται. Πώς να το δω. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος και εδώ άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία Ριμπέιρο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία της Επιτροπής Έμβι. Υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Που είναι ταυτόσιμη με την τροπολογία 14 της Επιτροπής ΕΒΗ. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχο, έλεγχος για την τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με ελάχιστη διαφορά. Δύο ψήφους. Τροπολογία 10. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Η 10 λέει καταπίπτει, λέει ο πρόεδρος. 9 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά το ελέγξουμε και ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 11. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Ίδια με την έμβη 9 υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Ποιο είναι υπέρ, λέει ο πρόεδρο, Εγκρίνεται. 15 και 16 μαζί υπέρ. Εγκρίνονται. 17 και 22. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. 18 υπέρ. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Εγκρίνεται. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία 20. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Εγκρίνεται. 23. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. Εκτός μικροφώνου τα σχόλια. Τροπολογία 23. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Εγκρίνεται. 25 υπέρ Εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 27 Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 28 και 29 υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. έρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Όντως απορρίπτονται. Τροπολογία 31. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 33, 34 και 38. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. 37. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 39 και 40 υπέρ. Εγκρίνονται. 41 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 42. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 42. Άρχεται η ψηφοφορία. 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 44 και έμβη για το 13 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 της ΕΜΒ. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. ΕΜΒ 8 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία της Επιτροπής Περιβάλλοντος, παριθμόν 8. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14 υπέρ, εγκρίνεται. Τροπολογία 15 της ΕΜΒ υπέρ, εγκρίνεται. Τροπολογία 350, ποιος είναι υπέρ. Κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 1 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Οπότε η 351 καταπίπτει. Αλλιώς θα έπρεπε να την ψηφίσουμε. Πάμε στην 369 τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 1 της έμβη υπέρ, εγκρίνεται. 370 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 371 υπέρ, κατά, Απορρίπτεται. 372. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 371. Πρώτα άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 372. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 375. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 της ΔΕΒ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. ΔΕΒ 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Αν επιμένετε. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την ΔΕΒ 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 386 του κύριου Άγγινου. υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 387 Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 396. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 397. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για την 397. Τέλος. Απορρίπτεται. Πάμε στις συμβαστικές τροπολογίες 4, 5, 6 και 7 που θα ψηφίσουμε μαζί. Ποιος είναι υπέρ, ή μάλλον ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Και πάμε στην τροπολογία 422. 422 της κυρίας Πετήρ. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για την 422 τροπολογία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 42 της ΕΜΒΗ. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την ΕΜΒΙ 42 Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 432. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 458 του κυρίου Βάιτς. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 459. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 463 της κυρίας Μαγκίνες. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 464. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Πολύ λυπάμαι. Πολύ λυπάμαι που καταψηφίσατε την τροπολογία μου. 465. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Α, διαβάσατε τι έλεγε η τροπολογία. Γιατί ε, ε, έχει σημαντική αιτιολόγηση. Διαβάστε την τροπολογία, γιατί ακολουθήσατε τους και ηγητές, αλλά δεν, δεν λάβατε υπόψη το συμφέρον των αγροτών. Πάμε στην 466 466 υπέρ εγκρίνεται. 468 ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Είναι διχασμένη αριστερά. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 469. Έχετε τώρα μία ευκαιρία να έρθετε στα συγκαλά σας. Ε, εγκρίνετε. Σας ευχαριστώ πολύ. 471. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Α, έτσι μπορεί να ξεχάσω το την προηγούμενη στεναχώρια. 64 MV υπέρ. Εγκρίνεται. 473. Ποιος είναι υπέρ. Κατά απορρίπτεται. MV34 υπέρ εγκρίνεται. 474 υπέρ εγκρίνεται. 475 υπέρ εγκρίνεται. 476 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 4 της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 481. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 482. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την 482. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 483. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 484. Υπέρ κατά απορρίπτεται. 486 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 486 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. 487 ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται. 488 υπέρ κατά απορρίπτεται. 489. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 489. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία 11 και πάμε στην τροπολογία 504. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 505. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 507. Υπέρ. Ή μάλλον πρώτα ηλεκτρονικός έλεγχος για την 505. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 507. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 508 υπέρ. Εγκρίνεται. MV63 υπέρ. Εγκρίνεται. 509 υπέρ. Κατά ηλεκτρονικό έλεγχο για την 509. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 510. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 512. Υπέρ. Εγκρίνεται. 513. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 514 υπέρ. Εγκρίνεται. 515 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 516 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 540. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 598. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Δεύε 19. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 542. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 543. Υπέρ. Εγκρίνεται. 548. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα την 551. Ποιος είναι υπέρ του κυρίου Μπέλτερ. Ποιος είναι υπέρ κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 551. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε τη συμβαστική 13. Ο κύριος Άγνιος ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, χάλασε το μηχάνημα της ψηφοφορίας εδώ μπροστά μου. Εγώ νόμιζα ότι άρχισε να ισχύει το Brexit. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 573 του κυρίου Κάρας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 573 η ψηφοφορία. Δεν είδα πώς ψηφίζει ο κύριος Βάιτς. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 578. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 579. Ποιος είναι υπέρ. κύριο Σάγνιο. Λυπάμαι που σας καθυστερώ. Αλλά η αγγλική διερμηνία συνεχίζει να λέει 470 κάτι και όχι 570 κάτι και με μπερδεύει. Λυπάμαι. Θα προσπαθήσω να μιλάω πιο καθαρά. 579. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Εγκρίνεται αλλά στο ελέγξουμε καλό κακό. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. «583 υπέρ εγκρίνεται, 584 υπέρ εγκρίνεται, 585 και 597 εγκρίνονται, 586 υπέρ εγκρίνεται. 589 υπέρ κατά απορρίπτεται. 591 υπέρ εγκρίνεται. 592 υπέρ κατά απορρίπτεται. 593 υπέρ κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 593 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με μία ψηφοδιαφορά. Λυπάμαι κυρία Νόιχλ. 595 και 596 υπέρ. Εγκρίνονται. 599 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 599 άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία 633. Πηδάμε δύο σελίδες. Μας αρέσει έτσι να τρέχουμε 633. Άρχι... Ποιος είναι υπέρ μάλλον. Ποιος είναι υπέρ της 633. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 633. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 637. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 634. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 636. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 636 άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 640. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και πάμε στην 657 τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 658. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 659 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 660 ή μάλλον πρώτα να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 659. Άρχεται η ψηφοφορία, μια και το ζητήσατε, για την 659 του κύριο Βάιτς. Τέλος ψηφοφορίας και απορρίπτεται. Τροπολογία 660. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 661. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 662. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 600... Μάλλον συμβαστική τροπολογία 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 688. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. χθες ε, κάναμε εξάσκηση. 695 695. Ποιος είναι υπέρ. Την 688 την εγκρίναμε ήδη, την ψηφίσαμε. Ή όχι. Την εγκρίναμε την 688. Την 695 δεν την ψηφίζουμε. Πάμε στην 689, στην επόμενη σελίδα. 689 της κυρίας Νόιχλου και άλλων. Κάντε Μπαχταραμπέλα Σάνι. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 689. Μικρόφωνο παρακαλώ. βλέπω 691 στο δικό μου κατάλογο το επόμενο. Εγκρίναμε την 687 και λέμε αν εγκριθεί πάμε κατευθείαν στην 689. Γι' αυτό περάσαμε στην επόμενη σελίδα. Στην 689 της κυρίας Νόιχλου και άλλων. Ποιος είναι υπέρ της 689 κατά Ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Εντάξει, έγινε μια ανταλλαγή απόψεων εκτός μικροφόνου. 690, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 694 του εισηγητού Ντόρφμαν. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 698. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 700. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 705 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 706 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 711 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 712 υπέρ Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 711. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μία ψηφοδιαφορά. 712 τώρα. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 713 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 713 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας και εγκρίνεται. 714. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας και απορρίπτεται. «716. Ποιος είναι υπέρ» «Κατά» «Ηλεκτρονικός έλεγχος». Και εδώ έρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 717 υπέρ κατά απορρίπτεται με την ίδια διαφορά 718 υπέρ εγκρίνεται 719 υπέρ κατά απορρίπτεται αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 719 ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία τέλος απορρίπτεται 720. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 721 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 722 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 17. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία 755. Ποιος είναι υπέρ της 755. Κατά. Απορρίπτεται. 760 και 761. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 763 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 758 Ποιο είναι υπέρ. 7.58. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Η κυρία Αγγιλέρα δεν σήκωσε το χεράκι. Έλεγχος για την 7.58. Άρχεται η ψηφοφορία. Τώρα. Αργά το θυμηθήκατε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 759. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πάμε στη συμβαστική τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 838. Της κυρίας Πετήρ. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 839. Υπέρ. Εγκρίνεται. 844. Ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται. 852 υπέρ. Μπούντα, ο κύριος Μπούντα δεν ψηφίζει. Εγκρίνεται παρόλα αυτά. 854. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 855 υπέρ. Εγκρίνεται. 857 και 858 Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται. Έχαμε πολλούς συντάκτες εδώ. 860. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 860. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος απορρίπτεται. Τροπολογία 865. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 868 υπέρ. Εγκρίνεται. 871 υπέρ. Εγκρίνεται. 875 υπέρ. Εγκρίνεται. 876 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 20. Άρχιτη ψηφοφορία. εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία 902. 902. Ποιος είναι υπέρ της 902. Υπέρ. Κατά. Μάλλον κάποιο λάθος κάνατε, γιατί έχουμε θετικό πρόσημα από το ΕΛΚ. Απορρίπτεται, φαίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 902, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Έχετε όλοι αρνητικό πρόσημο. Εδώ έχω μάρτυρα ότι το, ο δικός μου κατάλογος έχει θετικό πρόσημο και μάλιστα η ομάδα μου τον έδωσε το κατάλογο, το ΕΛΚ. «903. Ποιος είναι υπέρ» εγκρίνεται. 904 του κυρίου Βάιτς, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 907, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 911. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 913. Υπέρ. Εγκρίνεται. 916. Ε, υπέρ. κατά. Απορρίπτεται. 917. Υπέρ. Εγκρίνεται. 918. Υπέρ. Εγκρίνεται. 921. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 923 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 924 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 924. Άρχεται η ψηφοφορία. Μάλλον έχει εγκριθεί, μάλλον έχει απορριφθεί, συγγνώμη. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Και όντως απορρίπτεται. ήταν τροπολογία των αριστερών, της αριστερής πτέρυγας, αλλά ούτε η αριστερά δεν ψήφισε υπέρ. Πώς να το ερμηνεύσω αυτό. Τροπολογία 815. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε μαζί μάλλον παραλείψαμε την τροπολογία 914, δες γιάρ και άλλων, κατά Ψηφίζουμε την 914 των κυρίων δες και άλλων. Ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία αυτή. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Πάλι συγγνώμη που σας διακόπτω. Μόλις είπα... Όχι, τεχνικό λάθος που παραλήφθηκε από το κατάλογο και γι' αυτό σας είπα, το είπα στον εισηγητή. Και αν έχετε αφιβολίες ρωτήστε το για το περιεχόμενο. Κύριε Άγνιου, τρεις φορές είπα ότι κατά λάθος παραλήφθηκε, από τεχνικό λάθος παραλήφθηκε από τον κατάλογο ψηφοφορίας και το είπα στους συζητητές και στον ε, κύριο Ντόρφμαν. Εν πάση περιπτώσει, σημειώνω την παρατήρησή σας, αλλά το έχω επανειλημμένως ε, πει και σας ενημερώσει ότι είχε παραλυθεί κατά λάθο. Πάμε στις συμβαστικές τροπολογίες 21 και 22. Ψηφίζουμε μαζί ηλεκτρονικά. άρχιδη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Πάμε στην τροπολογία 959, τρεις σελίδες παρακάτω, Δες και άλλων. Ποιος είναι υπέρ της 959. Κατά. Εγκρίνεται ή θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Ηλεκτρονικός έλεγχος κατέτηση της κυρίας Αγγιλέρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 957 και 960. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. 961. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 966. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 973. Υπέρ. Εγκρίνεται. 981. Υπέρ. Για ποια τροπολογία ζητήσατε ηλεκτρονικό έλεγχο, κυρία Νόιχλ. 981 εγκρίνεται. 1012. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Τροπολογία 1004. Ποιος είναι υπέρ της 1004. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 1004 τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Η χιλιοστή τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 999. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 1009. Ποιος είναι υπέρ του κυρίου Χάσλινγκ. Κατά απορρίπτεται. Έμβη 16 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1010 του κυριο Βάιτς. Ποιος είναι υπέρ. Κατά Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 1010. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1011. Ποιος είναι υπέρ κατά. Απορρίπτεται. 1013. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 1014. Υπέρ εγκρίνεται. 1018 και 1019. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνονται. Συμβαστική τροπολογία 24. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος. Εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία 1047. Ποιος είναι υπέρ της 1047? Εγκρίνεται. 1058. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Η 56 καταπίπτει. 549. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 1048 υπέρ. Εγκρίνεται. 1049 υπέρ. Εγκρίνεται. 1053 υπέρ. Εγκρίνεται. 1055 υπέρ. Εγκρίνεται. 1059 υπέρ. Εγκρίνεται. 1061 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 1061. 1061 άρχεται η ψηφοφορία. Μα δεν ψηφίσατε υπέρ, τώρα το δηλώσατε. Τέλος ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 1063 Βάιτς υπέρ κατά απορρίπτεται. 1075 ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται. 1066 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 1066 άρχεται η ψηφοφορία τέλος Απορρίπτεται. 1067. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 1070 υπέρ. Εγκρίνεται. 1072 υπέρ. Εγκρίνεται. 1074 υπέρ. Εγκρίνεται. 1079 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1080 υπέρ κατά απορρίπτεται. 1081 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 1081 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. 1082 υπέρ κατά απορρίπτεται. 1083 και 1084. Ποιος είναι υπέρ, κατά απορρίπτονται. Ψηφίσουμε μαζί τις ε, συμβαστικές τροπολογίες 25 και 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνονται και πάμε στη 1098. 1098. Ποιος είναι υπέρ, κατά, Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 1098. Τέλος. Απορρίπτεται. 1101. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Δεν θέλετε κουπόνια για τα τρόφιμα. 1108 ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 1109 υπέρ, εγκρίνεται. 1116 και 1117 ποιος είναι υπέρ, εγκρίνονται. Συμβαστική 27 άρχεται η, η ψηφοφορία. εγκρίνεται και πάμε στην 1160. Ποιος είναι υπέρ, ο κύριο Βάιτς είναι ο συντάκτης, απορρίπτεται. 1150 και 1151, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνονται. 1154 και MV60, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνονται. MV61, υπέρ, εγκρίνεται. 1155 και 1161, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνονται. Συμβαστικές τροπολογίες 28, 29 και 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Πάμε στην 1189. 190 υπέρ. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 1190. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 1190. Τέλος ψηφοφορία. 31 και 32. Ψηφίζουμε μαζί. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνονται. Και πάμε στην 1211 του κυρίου Βάιτς. 1217 του κυρίου Βάιτς. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία. Εγκρίνεται. 1227. 1227. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 της Επιτροπής ή μάλλον Ηλεκτρονικός έλεγχος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10 της Επιτροπής Προϋπολογισμών υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τέλος. εγκρίνεται. 1257 της κυρίας Χάζεκαμπ. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 259. 1259. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 14. Ποιο είναι υπέρ, κατά, περ. Κατά, απορρίπτεται. 1261 του κυρίου Βάιτς υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Είναι τα ένα. Είναι τα 1, υπέρ, εγκρίνεται. Δεύ 3, 3, υπέρ, εγκρίνεται. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μικρή διαφορά. Ντεβε 12 τώρα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Τέλος. Απορρίπτεται. Ντεβε 13 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11 της Επιτροπής Προϋπολογισμών υπέρ. 5 υπέρ εγκρίνεται. 12, 69, 1269 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 1270 υπέρ, κατά, Ηλεκτρονική. Απορρίπτεται. 1271. Ποιος είναι υπέρ κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία για τη 1271. 52. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 1294 και ίντα 11. Ποιος είναι υπέρ. Κατά απορρίπτονται. Ίντα 4 υπέρ εγκρίνεται. Είναι το 14 υπέρ εγκρίνεται. Είναι το 15 υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 35. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται και πάμε στην... Ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται. 1289 υπέρ κατά απορρίπτεται. Δεύε 16 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 1291 υπέρ. Εγκρίνεται. Δεύε 18 υπέρ. Εγκρίνεται. 1292 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 1293 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 1296 υπέρ κατά απορρίπτεται. 12.98 υπέρ κατά απορρίπτεται. 12.99 υπέρ κατά απορρίπτεται. 1300 τροπολογία υπέρ εγκρίνεται. 1301 υπέρ κατά απορρίπτεται. 1302 υπέρ κατά απορρίπτεται. 1305 υπέρ κατά απορρίπτεται. 1306 υπέρ κατά απορρίπτεται. 1307 υπέρ κατά απορρίπτεται. 1308 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 13 της Επιτροπής Προϋπολογισμών υπέρ εγκρίνεται. Προϋπολογισμοί 14 υπέρ εγκρίνεται. Ίντα 7 υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 36. Άρχεται ψηφοφορία. εγκρίνεται. Τροπολογία 1319 υπέρ κατά απορρίπτεται. 1324 ποιος είναι υπέρ απορρίπτεται. 1322 υπέρ κατά Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 1322. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 1323. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 1325. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Σας περιμέναμε. Πάνω κάτω ο αντίχειρας. Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την 1325 του κυρίου Μέλο. Άρχεται η ψηφοφορία. Απ' την αρχή έπρεπε να το είχατε σηκώσει κύριε Αγγιλέρα. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Εγώ έχω θετικό πρόσημα. Δείχνει κατά η κυρία Αγγιλέρα, μπερδεύτηκα. 1326 υπέρ κατά, απορρίπτεται. 1327 υπέρ, εγκρίνεται. 1308 υπέρ, εγκρίνεται. 1329 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 1330 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. ΕΝΒΙΚ 62 υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 37 άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται και πάμε στην ΤΕΒΕ 8. Ποιος είναι υπέρ. Απορρίπτεται. ΤΕΒΕ 9 εγκρίνεται. ΤΕΒΕ 22 υπέρ εγκρίνεται. ΤΕΒΕ 23 υπέρ κατά απορρίπτεται. 924 24 υπέρ, κατά απορρίπτεται. 925 25 υπέρ, εγκρίνεται. 927 27 υπέρ, εγκρίνεται. 928 28 υπέρ, εγκρίνεται. 929 29 υπέρ, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 38. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 864. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 864. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβαστική 39. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία 517. Ποιος είναι υπέρ, υπέρ 517 Χάζεκαπ, υπέρ, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 40, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία 1297. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικό έλεγχο για την 1297. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορία. Απορρίπτεται και ψηφίζουμε μαζί τις συμβαστικές τροπολογίες 41 και 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνονται ψηφίζουμε μαζί τις τροπολογίες, συμβαστικές τροπολογίες 43, 44 και 45. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνονται. Συμβαστική τροπολογία Α. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 60. Εγκρίνεται. MV1 υπέρ. Εγκρίνεται. MVJ. Ε, εγκρίνεται. 76 της κυρίας Δελαέ. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία B. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 77. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία C. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία D. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος εγκρίνεται. Τροπολογία 115 και 116 παρόμοια. Ποιος είναι υπέρ εγκρίνονται. Συμβαστική τροπολογία Ι. E. ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 126 του κυρίου Βάιτς. Ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται. 127 και 128 υπέρ, εγκρίνονται. 130 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 131 υπέρ, εγκρίνεται. 132 και 133 υπέρ, εγκρίνονται. Συμβαστική τροπολογία F, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται και πάμε στην 134. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 134 άρχεται η ψηφοφορία. Της κυρία Σένερα και άλλων. Απορρίπτεται. 142 υπέρ του κυρίου Βάιτς. Κατά απορρίπτεται. 143-144. Ποιος είναι υπέρ μάλλον πρώτα ηλεκτρονικός έλεγχος για την 142. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 143 και 144. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. 145 υπέρ. Εγκρίνεται. 146 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 146. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Πάμε στην 151. Ποιος είναι υπέρ, κατά απορρίπτεται. 152, 153. Ποιος είναι υπέρ, εγκρίνονται. 154 υπέρ Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 154. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία G. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται και πάμε στην 173. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άρχεται ο ηλεκτρονικός έλεγχος για την 173. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ε, συμβαίνουν και αυτά. Απορρίπτεται. MVW. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται έμβη υπέρ εγκρίνεται έμβη υπέρ κατά απορρίπτεται ή μάλλον ηλεκτρονικός έλεγχος για την ΕΜΒΙΑΝ. άρχεται ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται 174 ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται 175 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία H Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 192 και 194 υπέρ κατά απορρίπτεται. Απορρίπτονται. 193 υπέρ κατά απορρίπτεται. 195 υπέρ κατά Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 195. άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Νόμιζα ότι έκανε λάθος ο κύριος Μπούντα. Κι εγώ μπερδεύτηκα. Πάμε στην 147. Ποιος είναι υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 197. Ποιος είναι υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 199 υπέρ. Κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 199 μάλλον επανάληψη ψηφοφορίας υπέρ κατά Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 199. Αυτό είναι άνω Μόνη Η κυρία Αγγιλέρα ψήφισε υπέρ της τροπολογίας της κυρίας Πετήρ. Απορρίπτεται. 201. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 202 υπέρ εγκρίνεται. Budget D, υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικό έλεγχος για την τροπολογία Δέλτα της Επιτροπής προπολογισμών. άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος, εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά. Συμβαστική τροπολογία I, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 219 των κυρίων Αντριού Ντενανότα Μπέλα. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 219. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 221. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. 224 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 224. Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 225. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία J. Άρχισε ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 241 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 241. Άρχισε η ψηφοφορία. Τέλος. απορρίπτεται. 246 και 247 υπέρ εγκρίνονται. 249 υπέρ εγκρίνεται. 250 υπέρ εγκρίνεται. 253 υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία κάπα Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. εγκρίνεται. Πάμε στην 58, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. τα ταφ υπέρ, εγκρίνεται. Έμβι α, εγκρίνεται. Έμβι κάπα, υπέρ, εγκρίνεται. 64, υπέρ, εγκρίνεται. 91, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. ιπέρ νι. υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 244 υπέρ εγκρίνεται. 245 υπέρ κατά απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 245. Αφού το ζητήσατε, τέλος ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Η MVM καταπίπτει. Όχι, όχι, δεν εγκρίθηκε η προηγούμενη, άρα θα πρέπει να ψηφίσουμε και την MVM υπέρ. MVM εγκρίνεται. Ας το επαναλάβουμε καλύτερα γιατί βιάστηκα. MVM. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας μη της Επιτροπής MV. Εγκρίνεται. Πάμε στην 267. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 100 72 του κυρίου Αρτουή, του Πρόεδρου της Επιτροπής Προϋπολογισμών. «172 του κυρίου Αρτουή». Απορρίπτεται. Νομίζω ψηφίσαμε από αυτή, λέει ο πρόεδρο. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα ξαναψηφίσουμε για αυτήν. Θα ψηφίσουμε τώρα για την τροπολογία L. Αυτό είναι λάθο στον κατάλογο για τον οποίο θέλω και να ζητήσω συγγνώμη. Τώρα έχουμε την τροπολογία, την ψηφορία για την συμβαστική L. Εγκρίθηκε Η 282 εγκρίθηκε, η 284 απορρίπτεται, NV 304 υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική N, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η συμβαστική Ο, ψηφίζουμε. 28 του κ. Βάιτς υπέρ παρακαλώ εγκρίνεται. Περνάμε στην συμβαστική π. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται συμβαστική Q. Ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 343 και ένβια αγιώτη υπέρ κατά αποχές ε, ε, ηλεκτρονική υπαλλήφθηση για 343 έκλεισε η ψηφοφορία εγκρίνεται Πάμε στην NVAK, υπέρ παρακαλώ, δεκτή. 3.46, κυρία Σράιρ, υπέρ, δεκτή. 3.47, υπέρ ΔΕΒΕ ΔΒ1 υπέρ κατά ηλεκτρονική επανελήθευση της Ein. 1 ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. Συμβιβαστική R. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Η S Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Επόμενο. Η τροπολογία 95 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβιβαστική T. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία εγκρίνεται, οπότε πάμε στην 960 U. Άρχεται η ψηφοφορία, συμβαστική τροπολογία U. Τέλος ψηφοφορίας. Ε, συμβαστική τροπολογία V για την αγροδοσοκομεία άρχεται η ψηφοφορία. εγκρίνεται και ψηφίζουμε το σύνολο της έκθεσης εγκρίνεται η έκθεση του κυρίου Ντόρφμαν Συγχαρητήρια κύριε Δορφόν και θερμά ευχαριστώ της αναγνώριση του έργου σας. Κύριε Ντόρφαν, έχετε το λόγο παρακαλώ. Να ευχαριστήσω όλους ε, τους ε, συνεργάτες μου σε αυτήν την έκθεση. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Αντριέ στην αρχή, ότι δεν μας παίρνει σοβαρά η Κομισιόν, οφείλεται σε μας το αν μας παίρνει σοβαρά ή όχι. Μα αλλιώς ε, έχουμε κι εμείς ε, τα μέσα ως ε, νομοθέτης να το κάνουμε. Και νομίζω ότι καταφέραμε ήδη με αυτήν την έκθεση να παρουσιάσουμε μια σαφή άποψη του Κοινοβουλίου με μια τη Μάγκη και τη Μαγδαλένα θα ήθελα να ευχαριστήσω και προσωπικά για το κολοσσιαίο έργο που επιτέλεσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Με... Δεν ζητά άλλο κανεί το λόγο, οπότε και πάλι θερμές ευχαριστίες προς τον εισηγητή μας και τους κοιόδη εισηγητές, τους συνεργάτες τους τη γραμματεία. Πάμε στο σημείο 6, τη διαφορετική ποιότητα των προϊόντων στην ενιαία αγορά εισηγητής ε, στα κράτη-μέλη και ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 11 του κυρίου Ροπέ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ. εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Στον κύριο Βιέγκας, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία. Εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία 66. Ποιος είναι υπέρ. Τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 112 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος είτε. οπότε ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης όπως έχει τροποποιηθεί με ονομαστική κλίση Άρα με μία αποχή και μία ψηφοκατά. Μήπως ο εισηγητής ο κύριος Νέκοφ θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Τη αποστολή πρώτα έχει το λόγο ο κύριο Αντρίε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για το, τον τρόπο της προετοιμασίας της επίσκεψης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την γραμματεία μας και το επιτελείο μας για την πολύ καλή διοργάνωση, αλλά καταρχήν μία πρώτη απορία για τη διάρκεια της αποστολής. Μετά θα περάσω στην ουσία. Η αποστολή θα πρέπει να προσέξουμε τους κανόνες και ίσως θα πρέπει να τροποποιήσουμε τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε δεν λέω να πηγαίνουμε δύο εβδομάδες και τη αποστολής έχω φιβολίες. Είναι κρίμα να πηγαίνουμε τόσο μακριά και να κρατάει τόσο λίγο αποστολή, ώστε να μην μπορούμε να αξιοποιούμε στο έπακρο την παραμονή μας εκεί. Ως προς το περιεχόμενο, έχω την ίδια αίσθηση με εσάς. Ήταν ε, υπερβολικά καλή η παρουσίαση ήταν ιδηλιακά θα έλεγα τα πάντα όπως μας τα παρουσίασαν. Και ίδιες ε, λέξεις, τα ίδια λόγια παντού, ίδιες καταστάσεις, παρά ήταν ε, εξειδανικευμένη παρουσίαση. Και παντού τις ίδιες απαντήσεις λάβαμε στις ερωτήσεις. Δεν λέω ότι ήταν κάπως ξύλινη γλώσσα, αλλά ήταν τέτοια η πολιτική ορθότητα και εξειδανίκευση που δημιουργούσαν κάποιες αμφιβολίες για την ουσία. Επίσης, ε, δεν μας καθησύχασε και πολύ αυτή η αποστολή. Γιατί εν ώψη των συμφωνιών με τη Μερκοσούρ διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν δύο κουλτούρες που βρίσκονται αντιμέτωπες. Έχουμε αφενός το θέμα της ε, σύγκρουσης συμφερόντων και έχουμε την ίδια ανάλυση της έννοιας της σύγκρουσης συμφερόντων και από ευρωπαϊκής πλευράς και από βραζιλιάνικης πλευράς. Ε, και στο Μάτο Γκρόσο που πήγαμε, στην πρώτη ε, συνάντηση που είχαμε με τον ε, Υπουργό Γεωργίας της Βραζιλίας. Ήταν πολύ καλή συνάντηση, αλλά είχαμε προβλήματα ως προς το θέμα των φυτικών καλλιεργειών. η σχέση της Βραζιλίας ε, με τις καλλιέργειες αραβοσίτου και σόγιας, γιατί έχουμε απέραντες εκτάσεις ε, γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου και σόγια στη Βραζιλία. Και μας είπαν οι Βραζιλιάνοι ότι παράγουν τέτοιους γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα γιατί πληρώνουν οι ευρωπαϊκές αγορές καλά. Και αν η μεγαλύτερη έτσι υπήρχε για τα συμβατικά προϊόντα θα, δεν θα κάναμε γενετικώς τροποποιημένα και για την αποψήλωση βλέπουμε ότι είναι σαφής η πρόσβαση. Γίνεται αποψήλωση των δασών, ε, το έδαφος είναι φτωχό, οπότε την αποψήλωση βλέπουμε ότι είναι σαφής η πρόσβαση. Γίνεται αποψήλωση των δασών, ε, το έδαφος είναι φτωχό, οπότε περνάμε σε καλλιέργεια γεννητικό τροποποιημένη σόγιας ή αραβόσιτου που δεν χρειάζονται πλούσια εδάφη και ε, φλωμώνουμε τις καλλιέργειες στη γλυφοσάτη. Δεν γίνεται φιδωλή χρήση τέτοιων ε, προϊόντων. Οπότε έχουμε σοβαρές ανησυχίες. Τώρα για το βόλιο κρέας που ήταν το μείζον ζήτημα. Ο κύριος Νταντά ίσως μίλησε αργότερα. Επισκεφθήκαμε κάποια σφαγεία και ε, ε, επισημάναμε το ζήτημα της ιχνηλασιμότητας. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες γιατί και εκεί υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες είδαμε ότι στην αλυσίδα του σφαγίου ε, τέθηκε θαυμάσια το ζήτημα της ιχνηλασιμότητας, γιατί μέσα στην αλυσίδα χάναμε τα ίχνη ε, του σφάγιου. Και θέσαμε σχετικές απορίες γιατί η ιχνηλασιμότητα αφορά την παρτίδα ολόκληρη. Οπότε τον αριθμό των ζώων που σφάζονται καθημερινά στο συγκεκριμένο σφαγείο. Αλλά είναι τεράστιες οι ποσότητες. Οπότε υπάρχουν κάποια κενά στην ιχνηλασιμότητα στα σφαγεία της Βραζιλίας. Και δεν έχουμε παρόμοια μοντέλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Βραζιλία. Εκεί είδαμε τις διαφορές που υπάρχουν και η εξασφάλιση της ε, χνηλασιμότητας σε τεράστιες παρτίδες 1.500 και ζώων που σφάζονται καθημερινά είναι αδύνατο. Φαντάζομαι και οι άλλοι συνάδελφοι θα το επισημάνουν. Αλλά για το θέμα αυτό, ε, τα όρια που είχαμε και στις φυτικές καλλιέργειες ε, και τις σχέσεις της Βραζιλίας προς τις γενοτικώς τροποποιημένες καλλιέργειες, αλλά και τα κενά που υπάρχουν στην ιχνηλασιμότητα, είδαμε κάποια πράγματα που δεν μπορούν να μας αφήνουν αδιάφορους ε, ως προς τις διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρμόσουμε στις μελλοντικέ μας συμβάσεις που θα έχουμε με τη Βραζιλία. Ο κύριος Κολομπιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για τον τρόπο που ε, οργανώσετε και διαχειριστήκατε αυτή την αποστολή και δώσατε το λόγο σε όλους τους βουλευτές και μάλιστα χωρίς περιορισμό και καταφέραμε να θέσουμε πολλές ερωτήσεις σε ό,τι αφορά τη διάρκεια, τη σύντομη διάρκεια της αποστολής, συμφωνώ με τον κύριο Αντρέα. Όταν πάμε στην άλλη άκρη του πλανήτη και έχουμε μόνο πέντε μέρες, εκ των οποίων οι δύο είναι το ταξίδι, νομίζω ότι η, ο κανόνας α, της τρίμερης παρανομής είναι πολύ περιοριστικός. Θα προτιμούσαμε να έχουμε πέντε μέρες επιτόπου για να κάνουμε μια πιο... Ουσιαστική έλεγχη ποιότητας, αυτό δεν νομίζω, δεν ισχύει, συμφωνώ με τον κύριο Νταντάν, αλλά θα ήθελα βέβαια και εγώ να... Στο βωμό των μεγάλων αυτών εμπορικών συμφωνιών, γιατί περί αυτού πρόκειται. Είναι τα εξηλαστήρια θύματα αυτών των συμφωνιών, η μικρομεσαία γεωργική κτηνοτρόφοι μας. Επίσης, η Βραζιλία ετοιμάζεται ε, να πουλήσει στην Ευρώπη και μάλιστα αυτοί που θέλουν να παράγουν κρέα για εξαγωγή προ την Ευρώπη με εξαγωγική προοπτική. Σε ό,τι αφορά τώρα την ποιότητα των προϊόντων. Είπαμε ότι γίνεται ε, εκτεταμένη χρήση της γλυφοσάτης και των γενετικών. αποτυπώματο άνθρακα για το κρέας τους. Γιατί αυτό ζητάμε και αυτό ετοιμάζονται να δώσουν. Είμαστε έτοιμοι να συνάψουμε τέτοια εμπορική συμφωνία. Πώς θα την αποτυπώματος άνθρακα για το κρέας τους. Γιατί αυτό ζητάμε και αυτό ετοιμάζονται να δώσουν. Είμαστε έτοιμοι να συνάψουμε τέτοια εμπορική συμφωνία. Πώ θα την πούν του μικρού καλλιεργητέ ή με μη κυβερνητικέ οργανώσει που θα μα μιλήσουν για τη γεωργική μεταρρύθμιση. Γιατί λόγω των μεγάλων ε, γεωκτημόνων έχουν στερηθεί οι μικροκτηματίες τη γη τους. Επίσης, τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τι γίνεται με την καταστολή στους ε, αγώνες των μικρο αγροτό στη Βρετανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ακούσαμε πολλά και ακούσαμε τη θεωρία της συνωμοσία ακόμη. Πάντως, μερικές φορές φαίνονταν ότι έχω κάνουμε μια έκθεση ελέγχου και όμως έχουν ε, και από την Επιτροπή πολλές επισκέψεις ε, ελέγχου και επιθεωρήσεων. Η δική μας επίσκεψη ε, προετοιμάστηκε από την Πρεσβεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με την Επιτροπή μας. Εγώ ρώτησα την Πρεσβεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάτι που φάνηκε κάπως μονόπλευρο, όπως είπαν οι συνάδελφοι. Γιατί δεν συναντήσαμε μη κυβερνητικέ οργανώσεις και με άλλους τομεί. Η απάντηση της πρεσβείας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν «Μα δεν μας το ζητήσατε». Εγώ έχω πολλές επαφές με μη κυβερνητικέ οργανώσεις και με άλλους τομείς και θα μπορούσα να τους είχα περιλάβει στην επίσκεψη, αλλά είχαμε και την πίεση του χρόνου. Η ε, επίσκεψη υπήρξε μια μονομέρεια ως προς του συνομιλητές μας. Ήταν όλοι από τη μία πλευρά. Ε, δεν είχαμε πιο ε, ευρύ φάσμα συνομιλητών. Επίσης, η ε, Βραζιλία είναι μια ηγετική χώρα ως προς την παραγωγή αλλά και ως προς την έρευνα της Γεωργίας και την κτηνοτροφία. Και μάλιστα πήγαμε σε ένα Ινστιτούτο που βρίσκεται στη πρώτη γραμμή τη έρευνα και έγινε μια παρουσίαση από το Διευθυντή που δείχνει πόσο προηγμένη είναι η έρευνα στην Βραζιλία για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Οπότε δεν πρωτοστατεί μόνο στην παραγωγή αλλά και στην έρευνα η χώρα αυτή. Κάτι που διαπιστώσαμε και που δεν ακούσαμε ακόμη τους συναδέλφους είναι ότι ο Υπουργός ε, είπε κατηγορηματικά ότι ε, η συμφωνία Μερκοσούρ ε, χωρίς το κεφάλαιο της Γεωργίας δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στα, στον αμπελονικό τομέα και σε άλλους κλάδους, οπότε σίγουρα και για αυτούς είναι προβληματικό το θέμα της συμπερίληψης όχι της γεωργίας. Γιατί αυτοί ενδιαφέρονται να ε, πουλήσουν κρέας, να εξαγάγουν κρέας. Και έχουν συμφέρον και ενδιαφέρον να, να βρουν κάποια κοινά σημεία επαφή στη διαπραγμάτευση. Κάτι άλλο που έκανε η Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, δύο λεπτά μίλησα, άλλοι συνάδελφοι μίλησαν έξι. Ε, όταν μιλήσαμε για την Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωρίζουν το Μερκοσούρ, ε, στις Συμφωνίες Ελεύθερων Συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε δεν το γνώριζαν καν. Γνώριζαν για το Μερκοσούρ, γνώριζαν για άλλες επιμέρους συμφωνίες, αλλά ότι ε, γίνονταν λόγος διαπραγματεύσεις Συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαίνεται να το γνώριζαν. Επίσης, το θέμα του κλίματος και της βιοπικιλότητας. Η Βραζιλία έχει ένα πανίσχυρο Ινστιτούτο, το ΙΜΠΑΜΙ, που έχει και ενεκτικές εξουσίες. Και μάλιστα η χώρα αυτή δεσμεύθηκε υπέρ της προστασίας της βιοπικιλότητας και της καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών. Οπότε σίγουρα και η Γεωργία και η δασοκομεία τους λαμβάνει υπόψη αυτό το θέμα. Και η ρητορική της Βραζιλίας είναι μια ρητορική που θεσμικά τουλάχιστον ε, λέει ότι η Βραζιλία έχει δυνατότητα να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση της προάσπισης της βιοποικιλότητας. Επίσης, έχουμε πολλά κοινά σημεία με τη Βραζιλία και ο λαός, ο βραζιλιάνικος λαός είναι πολύ συμπαθής. Γι' αυτό μερικές φορές η εριστική συμπεριφορά κάποιων συναδέλφων στην αποστολή ήταν δυσάρεστη. Μερικές φορές έδειξαν την φύση τους ως Ευρωπαίοι. Φυσικά υπήρξαν κάποια κενά στη συζήτηση υπάρχουν κάποια προβλήματα κακής μεταχείρισης των εργαζομένων που μοιάζουν ε, σαν να είναι πραγματικά ε, υποδουλωμένοι και όντως έχουν πολύ χαμηλό εργατικό κόστος. Πάντως και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε διαφθορά, έχουμε και εμείς πολλές αχίλες πτέρνες, δεν είμαστε άψογοι, δεν έχουμε δικαίωμα λοιπόν να δίνουμε μαθήματα σε άλλους και το δικαστικό σύστημα στη Βραζιλία είναι πολύ ισχυρό και μάλιστα προσπαθεί να επιλύσει αυτή τη στιγμή αυτό το πρόβλημα. Αντίστοιχε προσπάθειε κάνουμε και εμεί να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά κύριε Πρόεδρε, ήθελα να δώσω και τη δική μου εκδοχή και την άλλη άποψη που μέχρι στιγμής δεν ακούστηκε στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ε, παρατράβηξε η συζήτηση ε, μην ξεχνάτε ότι ακολουθεί η συνεδρία των συντονιστών. Οι τη μακρηγόρησαν. Οι υπόλοιποι παρακαλώ ε, να είναι πολύ πιο σύντομοι και απλώ να υποβάλουν ερωτήσει αν υπάρχουν. Ο κύριος Ντες ήδη υποσχέθηκε ότι θα μιλήσει δύο λεπτά. Ένα λεπτό παρακαλώ κύριε Ντες. Ευχαριστώ. Ε, φιλανθρωπική στην Βαβαρία ε, Έχουμε συγκεντρώσει μέχρι και 80.000 περίπου ευρώ ως ε, με τη μορφή δωρεών ε, διανυκτερεύσει ε, και πληρώσαμε 3.000 ευρώ. Πρέπει λοιπόν να το συζητήσουμε εδώ τι γίνεται, πόσο κοστίζει σε εμά ένα ταξίδι. Ούτε... αυτό, αυτά είχα να πω, πέρασε και το λεπτό μου. Τα έκανα, εάν είχα πάει, θα ήταν ο βαθμός της χρήσης αντιβιωτικών στα λέει καθόλου σοβαρά στην ε, Βραζιλία. Σας ευχαριστώ κύριε Φλάνακα. Σας ευχαριστώ ούτε εγώ πήγα στην αποστολή, διάβασα την έκθεση. Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι η εντύπωση να δίνεται η εντύπωση ότι το σπίτι κάποιου είναι ανάκτορο. Και εδώ πέρα λοιπόν το, το σαλόνι μας, έδωξε, μας έδειξαν. Αν ήταν αυτό το σαλόνι τους, ας φανταστούμε τα υπόλοιπα. Μας λέει ο κύριος Νταντών ότι εδώ πέρα δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η χνηλασιμότητα. Αυτό και είναι διατεθειμένοι να κάνουν τα πάντα και να πούν τα πάντα. Και μετά ο κύριος Νίκολσον είπε ότι ε, σας είπαν τα ίδια πράγματα πριν από 10 χρόνια και μετά από 10 χρόνια δεν έχει αλλάξει τίποτα. Επίσης ο κύριος Νίκολσον είπε αγρότες μας. Εγώ είχα κάνει μια εκδήλωση στην ε, Ιρλανδία για την βιολογική κτηνοτροφία. Επισκεφτήκαμε αγροκτήματα σε περιοχές όπου προστατεύεται η φύση και είχαν ελάχιστο αντίκτυπο